Ροβάνα Πλούμ μου ανέφερε την, το διορισμό της στην κυβέρνηση της Ρουμανίας. Βάσει του άρθρου για την εκλογή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κοινοβούλιο ε, διαπιστώνει την χειρία της θέσης της κυρίας Ροβάνα Πλάμπ. Και θα ήθελα να συγχαρώ ε, την κυρία Πλάμπ για την εκλογή της και θα μπορούσε να τα διαβιβάσει αυτά τα συγχαρητήρια ο κύριος ε, Σφόμποντα. Επίσης, ε, η, εντολή της κυρίας Λάγκ